την τροποποίηση της ημερησίας διατάξεως. Όταν λοιπόν θα φτάσει η συζήτηση στο σημείο το οποίο ασχολείται με την απαλλαγή θα σας καλέσω να κάνετε τις σχετικές σας παρατηρήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Περνούμε λοιπόν στην ημερήσια διάταξη έτσι όπως, ε, ε, όπως ορίστηκε από, την, ε, από τους Προέδρους των ομάδων. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις τροποποίησης της ημερησίας διατάξεως. Τετάρτη 2 Απριλίου. Η κοινή συζήτηση για την κοινή εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας μεταφέρεται για την 5η το πρωί αντικαθίσταται δε από την έκθεση Wilmot ε, για τις κλινικές δοκιμές και θα ακολουθηθεί από κοινή συζήτηση για τις ηλεκτρονικές ε, επικοινωνίες. Δεύτερον, η σύσταση της κυρίας ε, Μούνιτ Ουρκίθα. Ε, έχει αποσυρθεί από την ημερήσια διάταξη η δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής είπα της εκπροσώπου της Ένωσης για την κατάσταση στο Ιράν θα γίνει την Πέμπτη το πρωί μετά την κοινή συζήτηση για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας. Η δε συζήτηση θα ολοκληρωθεί με ψήφισμα της ΑΦΕΤ. Τρίτον, τα ακόλουθα θα ε, θέματα συμπληρώνουν την ημερήσια διάρκεια της σήμερα. Έκθεση Wilmot για τις κλινικές δοκιμές, έκθεση Κλέβα Κέκου σχετικά με τι μητρικέ εταιρείε. Τέταρτη ανακοίνωση. Τα ακόλουθα θέματα μετατίθενται από τις, σημερινέ τις σημερινές ψηφοφορίες της Οι δύο εκθέσεις Καρύμ σχετικά με τις υποχρεωτικές, ελέγχου. υποχρεωτικούς ελέγχους. Ε, καθώς επίσης και η έκθεση Ντονζόν ε, θα ψηφιστούν αύριο. Η έκθεση Γκαρίγκα Πολέντο σχετικά ε, με την πρόβλεψη εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2015, καθώς επίσης και η έκθεση Κασπαρή για τις δημόσιες προμήθειες βγαίνουν, αφαιρούνται από τη μερίσια διάταξη. Πέμπτον, η πρόταση της χειρισίστας της κυρίας Όμεν Ρόιτεν σχετικά με την κοινοτικότητα των εργαζομένων αφαιρείται και αντικαθίσταται από την έκθεση Ζαλεύσκη σχετικά με μείωση και ενδεχόμενη απαλυφή των τελωνιακών δασμών προϊόντων που έρχονται από την Ουκρανία. 5η-3 Απριλίου. Τα ακόλουθα θέματα θα συζητηθούν την 5η το πρωί. Κοινή συζήτηση για την κοινή πολιτική ασφάλεια και εξωτερική πολιτική. Ε, δήλωση τη Αντιπροέδρου τη Επιτροπή ε, ΥΠΑ εκπροσώπου ε, για το Ιράν και έκθεση Φιέλν για, ε, για προϊόντα διπλής χρήσης. Οι ψηφοφορίες Δελκαστίγιο ε, και Ουλσκοκ ε, θα παραμείνουν και θα λάβουν χώρα την Πέμπτη το πρωί. Αυτές είναι οι αποφάσεις που έλαβε η διάσκεψη των Προέδρων. Έχετε κάποιες παρατηρήσεις ή σχόλια. Όχι από ό,τι φαίνεται, επομένως αυτές οι τροποποιήσεις έχουν εγκριθεί και επομένως ορίζεται με αυτόν τον τρόπο το χρονοδιάγραμμα των εργασιών μας. Ας ξεκινήσουμε τώρα τη συζήτηση των διαφόρων εκθέσεων. Θα ξεκινήσουμε με την έκθεση του κυρίου Βίλμοτ σχετικά με τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων για χρήση σε ανθρώπους, για ανθρώπινη χρήση. Παρακαλώ πολύ. Βίλμοτ. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδης συζητητές για τη θαυμάσια στήριξη και συνεργασία. Μαζί καταφέραμε να επιτύχουμε πολλά για το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ και την Λιθανική Προεδρία